σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση και να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι, έχω διάφορες ανακοινώσεις. Μετά την τελευταία σύνοδό μας ε, που έληξε στις 7 Ιουλίου, στις 7 Ιουλίου ε, ε εγκρίθηκαν και τα πρακτικά. Δεν έχετε σχόλια, βλέπω. Όχι, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Βάσει του άρθρου 211 παράγραφος